Η ημερήσια διάταξη ε, μας επιβάλλει την εξέταση της έκθεσης Κοφεράτη σχετικά με την πρόταση οδηγίας ε, για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσης ενεργού συμμετοχή των μετόχων και μια στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω